Good afternoon, colleagues. Καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εβδομάδα πριν από τι διακοπέ. Σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε τρεις εκθέσει και αύριο άλλε πέντε. Οπότε το Σεπτέμβριο θα πάει κάτι από εμά στην Ολομέλεια θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα, πρόταση κανονισμού για το προενταξιακό μέσο αρρωγής, η έκθεση Κριστιαν Διγέννη. Και ξεκινώ αμέσως επειδή έχουμε πολλές ψηφοφορίες σήμερα. Άρθρο 1, τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προπολογισμό 16. Τμήμα 1. Είναι σε δύο τμήματα. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. «119 υπέρ». Όχι, συγγνώμη. 121. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 128 υπέρ. Εκατόν είκοσι 128. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 και ρέτζι 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 και employment 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμός 16 στο δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Θέλετε έλεγχο για την 16, δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται πράγματι. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προϋπολογισμός 16 το τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. η γραμματεία μου λέει ότι εκπίπτει η 16 τρίτο τμήμα διότι εγκρίναμε τη 133. 30 του εισηγητή υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. τα 8 κατά άποχες Είναι τα 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές. Χρειαζόμαστε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο στην 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1.36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Απασχόληση 19. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσχόληση 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 και 138 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 140 και έτσι 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Απασχόληση 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ρέτσι 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 και 127 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 142 υπέρ κατά αποχές. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 142. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 143 και ρέτζι 12 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 34 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Budget, υπολογισμός, 16 τέταρτο τμήμα υπέρ κατά Υπέρ και πάλι. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. 16 προϋπολογισμών. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το τέταρτο τμήμα. Πέρασε. 21 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται, πάση Απασχόλη 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 12. Όχι, όχι δεν είναι. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 145 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 146 και απασχόληση 25 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 147. Πέρας. Εγκρίνεται. Τριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απασχόληση 27 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές <coughs> κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο Πέρας. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ όμως σηκώντε τα χέρια σας για να κερδίσουμε και χρόνο. Είναι τα 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Είναι τα 13 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά μονάχα. Προπολογισμό 17. Τρίτο τμήμα μονάχα, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 38 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Απασχόληση 28. Όχι, εκπίπτει. 39 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. 51 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 41 έχει αποσυρθεί. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μην τα 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 155 ηλεκτρονικά Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 και budget 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμός Ρέτζι 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο στην 159 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας απορρίπτεται Ρέτσι 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 και 162 ίδιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται απασχόλησης 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμού 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Προπολογισμού 20. Άλλο ένα, τώρα εντάξει. Απορρίπτεται. Πράγματι. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμού 21 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την τροπολογία 21 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Πέρα τις ψηφοφορίες απορρίφθηκε. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμών 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απασχόληση 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 και απασχόληση 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 25. Μόνο το πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντα 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμών, όχι, καταπίπτουν. 58, τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Κανείς αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 178 και απασχόληση 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 36 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Το ΕΛΚ δεν δείχνει. Απασχόλησης λοιπόν, τροπολογία 36. Πέρυσι ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προπολογισμό 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμό 27 υπέρ. Όχι. Ρέγγι 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. τα 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 185 και ρέγγι 21 που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμών. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Ελέγχουμε 186 τροπολογία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. 27 υπέρ, 19 κατά. 28 προπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 τώρα. 72 διορθώνω ο πρόεδρος. 72 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 38 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προπολ... 195 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προπολογισμό 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 197 και απασχόληση 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ρέγγι 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202. Ποιοι είναι κατά τις 202 παρακαλώ. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε παρακαλώ για 202. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα για μένα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ναι, απορρίπτεται. Απορρίπτεται σαφώς. Είναι ξεκάθαρο ότι απορρίπτεται. Κύριε Κορνέλη, συνείδατε. Το προσπάθησε έτσι, δεν έχετε παράπονο. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προπολογισμό 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε προπολογισμό 3. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 3 της Επιτροπής Προπολογισμών. Πέρα της προφορίας. Απορρίπτεται πράγματι. 25 κατά και 19 υπέρ. Προπολογισμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Όπως και πριν. Απορρίπτεται. Προπολογισμών 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 6. Υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Απασχόληση αριθμό 1 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 82. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπόλιο 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 82. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 80. 2. Απορρίφθηκε. 22 ψήφοι κατά, 20 υπέρ. 2 δεν ψήφισαν. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα 3 του συγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 89. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Ίντα 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόλησης 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογισμών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ανεπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμών 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12. Όχι, λάθος. Διορθώνει ο πρόεδρος. Ρέγγι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προπολογισμό 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απασχόληση 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, α, όχι 18 διορθώνω ο πρόεδρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 και 112 που είναι ίδιες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Προπολογισμόν ένα δεν την ψηφίζουμε. Και έτσι τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Δεν έχει τελική ψηφοφορία. Πάμε στην επόμενη έκθεση που ψηφίζουμε let's. You take your voting list. Okay. Yeah. Thanks so much. Mr. Vigenin. Uh, Mr. Vigenin wants the floor. Two seconds. Mr. Vigenin has the floor. Yes. Okay. Thank you. Very briefly, I would like to sincerely thank the shadows for... Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους εισηγητές από τις διάφορες επιτροπές και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ψήφισαν την έκθεση σε αυτή τη φάση μετά από διαπραγματεύσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να κάνουμε τώρα μια, ψηφοφορία για την έναξη των άτυπων διαθεσμικών διαπραγματεύσεων σε σχέση με τις τροπολογίες. Πρόκειται για την εντολή σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Έχουν γίνει δεκτές. Έχει γίνει δεκτή η εντολή μάλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στην έκθεση για το μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κούκαν. Έχετε να πείτε κάτι κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να κάνω εγώ τελικά σχόλια, αλλά για να πάνε καλά τα εκλογικά μας, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους σχετικά με την προφορική τροπολογία την οποία καταθέτω μετά από συμφωνία ανάμεσα στον εισηγητή και του σκιώδης. Υπάρχουν τέσσερις προφορικές μάλλον τροπολογίες η μία αφορά, η μία είναι η συμβιβαστική 1, η οποία στο άρθρο 1 παράγραφο 1 αναφέρεται στη δημιουργία ενός χώρου σταθερότητας, ευημερίας και σταθερότητας και ειρήνης. Προσθέτουμε τη λέξη ειρήνη. Έχω επίσης την τροπολογία υπαρίθμου 0 σχετικά με την 2.13 την τροπολογία 2.13. Είχαμε ήδη συμφωνήσει ότι θα επανισάγουμε την εξή φράση «Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των χωρών και των συνεργαζομένων χωρών θα ποικίλουν οι ενισχύσεις αυτές ανάλογα με την προσπάθεια που γίνεται για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα πάντα στο 1 για την 2.19 υπάρχει μια νέα παράγραφος 1α για την αφαίρεση μίας λέξης, της λέξης enhance, βελτιώνω. για την τροπολογία Wiggening 85 πρόκειται για μια συμβιβαστική τροπολογία η οποία λέει το εξής έτσι ώστε να διευκολύνουμε την εφαρμογή της αρχής more for more και τη σωστή κατανομή των πιστώσεων θα θα χαρακτηριστούν εντατικές μορφές ενίσχυσης ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες αποδεικνύουν συγκεκριμένα βήματα προόδου για την εγκαθίδρυση, ενίσχυση της δημοκρατίας και την εφαρμογή των συμπεφωνημένων στόχων. Ε, Ζάλα. Κύριε Ζάλα, σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία με 123 προσθέτω μέσα σε αγγείλη το ότι η Τουρκία είναι Τουρκία ως υποψήφια χώρα μέσα στις αγγίλες. Μα μπορούμε να κάνουμε προφορικές τροπολογίες όταν ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Αν το κάνουμε αυτό συνέχεια θα ψηφίζουμε μόνο το προφορικέ τροπολογίε. παρατηρεί ο κύριο Μπροκ. Α ξεκινήσουμε την ψηφοφορία και θα έρθουμε αργότερα στην προφορική τροπολογία. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχέ. Δεκτή. Η 27 εκπίπτει. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εκπίπτει. Απορρίπτεται μάλλον. Είναι τα 10 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 145, 146, 147 ταυτόσιμες είναι καλό να σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο λέει ο πρόεδρος και να χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια διατύπωση τους βοηθεί και το Άγιο Πνεύμα ενδεχομένω. ψήφι υπέρ κατά Ας Πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκτές. Περιφερειακή 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Προπολογισμό 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 156. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προπολογισμή 11. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Κατά μάλλον. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προϋπολογισμή 12 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 10 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ίντα 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Dev 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 166. Τη κυρία Γκάλ και Ρέτζι 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ίντα 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρασε. Oh. 170 in favor. υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 18 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Budget 14 υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα, νομίζω ότι είναι υπέρ αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ψηφίσατε όλοι. 26 υπέρ, 20 κατά δεκτή. Ήτρο 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φτάνουμε τώρα στην 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 και προϋπολογισμός 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πολιτισμός 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, η γυναικών 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πολιτισμός 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ίντε 16 υπέρ κατά αποχές Δεν ξέρω εδώ πώς θα έπρεπε να, έπρεπε να είχαμε μιλήσει πρώτα με την κυρία Πακ. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Απασχόληση 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πολιτισμός 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέγγι 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι ε, ε, ή μάλλον 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προϋπολογισμός 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 του εισηγητή. Για μια στιγμή διακόπτει ο πρόεδρος. Πολιτισμός 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προϋπολογισμός 19 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 19 της Επιτροπής Προϋπολογισμών ψηφίζεται πέρα στις ψηφοφορίες 27 υπέρ 18 κατά γυναικών 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 203 υπέρ κατά αποχές δεκτή 204 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 204. «27 υπέρ 18 κατά, προϋπολογισμός 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». Είναι τα 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήτρε 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39. Πέρα της ψηφοφορίας. 38 οκτώ κατά. Να θυμίσω στα μέλη να σηκώνουν τα χέρια τους κάπου κάπου. 205 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 206 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 209, 210, 11. είναι μια κοινότηση ε, πνεύματος και εργασίας, οι τρεις η ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 212 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 213 με προφορική τροποποίηση από τον εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 219 με προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 ε, γυναικών. ...18 γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.28 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές άρχεται ηλεκτρονικός έλεγχος Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σαράντα πέντε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 230 υπέρ κατά απορρίπτεται. Δύο τριάντα ένα, δύο τριάντα δύο, δύο τριάντα τρία και τα λοιπά. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Προϋπο, ε, κουλτούρα 24, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Για την ΔΕΒΕ 15. Πέρας απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμό 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.35 κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είτε 30 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είτε 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέγγι 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Λοιπόν, πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας, όμως δεν, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Αν είσαστε πολύ κουρασμένοι, παρόλα αυτά κάντε μια προσπάθεια. Μήπως πρέπει να μας φέρουν καφέ. Τι γίνεται, γιατί δεν μας έχουν φέρει καφέ, λέει ο πρόεδρος. Ποια ήταν η τροπολογία τώρα που ψηφίσαμε. Λοιπόν, 48 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 239 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 προϋπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 του εισαγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτερ 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι ομάδες εργασίες 241, 242, 243 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 εκπίπτει. 31 προϋπολογισμοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 του εισηγητή κατά αποχές εγκρίνεται. 52 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50, 53 προηγουμένως. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές δεκτή, 20 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ήτρε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, προϋπολογισμή 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμοί 35 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 56 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 22 γυναικών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 57 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 προϋπολογισμών εκπίπτει. 24 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.49 μέχρι 2.51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2, 53 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτούρα 25 υπέρ κατά απο, απορρίπτεται Ρέτζι 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.55 όχι εκπίπτει. Εκπίπτει και 38 και 22. 2.56 και ρέγγι 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέτζι 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέτζι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέτζι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 259, 260, 261. Υπέρ. Κατά αποχές. Ρέγγι 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφεται 262 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφεται 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.64 εκπίπτει. Ρέγγι 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 29 υπέρ. Κατά δεκτή. Ρέγγι 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 62 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2.66 εκπίπτει. 63 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ρέτζι εκπίπτει 65 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προϋπολογισμή 37 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2,70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 22 υπέρ κατά. Πάλι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά. Έλεγχος. Πέρασε. 21-27 απορρίπτεται. Γυναίκε 25. Ψήφι υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. Ίντα 25, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 του εισηγητή, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Ήτρε 39, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 33, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 273, 274 κουλτούρα 27, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 και 39 προϋπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 275 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 276 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 69 και 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προπολογισμού 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 προπολογισμοί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΔΒ1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 κατά αποχές Α, όχι μόνο το μία φράση πρέπει να ψηφίσουμε. Έλεγχο στη δύο καταρχήν. Πέρας ψηφοφορίες. Όποιος ζητάει έλεγχο, ίσως ήξερε εκ των προτέρων τι αποτέλεσμα θα βγει. Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Εβδομήντα τρία μόνο ψηφίσουμε τη φράση through an adequate mechanism. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Στην 74 μόνο το country specific. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κάνουμε έλεγχο μάλλον. Πέρας. Δεκτή η 74. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο γυναικών υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρεγγι 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 3 υπέρ. Κατά αποχές αποχές απορρίπτεται, γυναίκες 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ κατά αποχές, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21-26 απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Επτά του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά απόχε, δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 και ρέτζι 2 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές. Πάλι 104 υπέρ κατά απορρίπτεται. 9 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τεβε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 3 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έχουν εκπέσει Πολιτισμός 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 11 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. ρέτσι 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 5. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ή 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 13 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 14 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτούρα 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κουλτούρα 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτούρα 7. Εκπίπτει. Ή 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κύριε Τσάλα, θέλετε να πείτε κάτι εδώ. Κύριε Τσάλα. Έχει φύγει ο κύριος Τσάλα. Προφορική τροπολογία ήταν. Να το ξαναπώ. Ναι, ναι. Ξέρετε τι λέει η τροπολογία μου το πρότεινα, το ανέφερα στην αρχή της ψηφοφορίας. Τον Τσά το ξέρει, αλλά εγώ έχω ξεχάσει, λέει ο πρόεδρος. πως μπορείτε να μας καταπείτε. Στην τροπολογία 123, μια αλλαγή που μιλάει για Τουρκία και ε, Ρωσία. Θέλω να αλλάξω την Τουρκία ως υποψήφια χώρα μέσα στις αγκύλες. West. Ψήφι υπέρ της 123 με αυτή την τροποποίηση. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. Πέρας. «23-25 απερίφθη». Πού ήμασταν? 124 και ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι τα 6 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτουν όλες αυτές. Πάμε στην 130 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Επτά των προϋπολογισμών. Επτά προϋπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές 131 υπέρ κατά πρέπει να κάνουμε έλεγχο πέρας ψηφοφορίας. Κύριε Σαρσβόλσκι, βλέπετε δεν μπορεί κανείς να υποδείσει την τροπολογία σας να περάσει. Εγκρίνεται. Πολιτισμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβέστη 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 γυναικών υπέρ. Κατά από έλεγχος. Πέρας. 21 με 27 αποδείπτω. 6 απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 απασχόλησης υπέρ. Πούντινε, πούντιν, πούντιν. Υπέρ της 7 απασχόλησης, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτούρα 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24, 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Κουλτούρα 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας για την κουλτούρα 16. 22-26 απορρίπτεται. 17 κουλτούρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε κατά συνέπεια στην εντολή διαπραγμάτευσης. Ποιο μα δίνει εντολή για να διαπραγματευτούμε επί αυτή τη βάση η ψήφι υπέρ, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά όμω. Ηλεκτρονικά. Πέρα τη προφορία. υπέρ, καμία ψηφο κατά και τέσσερι αποχέ. Ούτω απεφασίστη. Κύριε Κούκαν, Είναι πραγματικά ισχυρή η εντολή που σας υποστηρίζει και αυτό είναι και επικίνδυνο κιόλας. Και τώρα η ψηφοφορία της έκθεσης για το εργαλείο εταιρικής σχέσης. Κύριε Μάουρου, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1-1-4. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. στις ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ένα, δύο, τρία. Ψήφου. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μαύρο σχετικά για την 123. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, να πω ότι θα καταψηφίσω την προφορική τροπολογία. Ψήφ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τρία, Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τα 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφήστε τον κύριο Μάουρο ήσυχο σας παρακαλώ να ψηφίσει με την ησυχία του, χωρίς περισπασμούς. Πού ήμασταν? Στην 26. Ηλεκτρικός έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε 21-22 αλλά απορρίπτεται. Δεν ήθελα να πω τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια των ψηφοφοριών, αλλά θα ήθελα να μας δίνετε και κάποιες ε, ψηφοφορίες, κάποιες πληροφορίες για το πόσοι είναι οι πράσινοι στην αίθουσα τώρα. Από ό,τι ξέρω έχουν έξι ψήφους, αλλά μου φαίνεται ότι ψηφίσουν 7 πράσινοι. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά και πρέπει να μας πει η γραμματεία πόσες ψήφους έχουν οι πράσινοι σε αυτή την επιτροπή. Μπορεί να το επιβεβαιώσει η γραμματεία ότι είναι ακριβώς όσοι πρέπει να είναι. πρέπει να κάνουμε προσπάθειε στι επόμενε εκλογέ εκλογές να τους περάσουμε, γιατί έχουν 7 τελικά έδρες στην, στην Επιτροπή μας, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, απορρίφθηκε 26, 21, 22 όπω σα είπα. ΔΒΗ 12 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορριπτεύεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 134 κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα κατά αποχές απορρίπτωται. Δεύτερο τμήμα κατά αποχές απορρίπτωται. ΔΕΒΕ 14 υπέρ έλεγχος προηγουμένως στο δεύτερο τμήμα της 134. Πέρας. 21-23 απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμοί 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές Έλεγχος για την 142. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-22 ισοψηφία, αλλά απορρίπτεται. 1-43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύε 18 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμοί 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 147 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 150 μέχρι 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 159 και 33 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ή τα 22. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι, 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 προϋπολογισμοί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προϋπολογισμή 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 εκπίπτει, εκπίπτει, εκπίπτει. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμού 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται, συγγνώμη. Υπέρ για 18 προπολογισμών. Πάλι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 του εισηγητή. Κατά από... Δεκτή, 19 προπολογισμοί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 του εισηγητή 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ...39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι 30 εκπίπτει, 41 του εισηγητή 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 εκπίπτει. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 22 υπέρ κατά απόχέ δεκτή. 43 του εισηγητή υπέρ κατά απόχέ δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήντα 32 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 45 του εισηγητή και τα 33 Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τρία προϋπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμή τέσσερα. Τέσσερα και πέντε μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Είναι τα ένα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρα ένα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκ... απορρίπτεται. Είτε 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 3-2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 12 σε 3 κομμάτια. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Έλεγχος. Για το τρίτο τμήμα. Ωραία. Πέρας φοφορίας. Πέντε δεν ξύπνησαν για να ψηφίσουν. Πέρα ψηφοφορίας. 24 προς 17 γίνεται δεκτή. Τροπολογία 5. 6 και 7 μαζί. 5, 6 και 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Συμβαστική 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα η ίδια κατά αποχές μάλιστα δεκτό. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 98 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Πάμε στην ε, ΔΕΒΕ1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καλησπέρας Στον έλεγχο. 20 με 21. Απορρίπτεται. 100 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Είναι τα 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 5 Πέρας. «21-20 γίνεται δεκτή. Ήτρε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. τα 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προϋπολογισμός 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕ3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕ4 σε 3 φέτες πρώτο τμήμα κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τρεπτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ όλες μαζί 105 μέχρι 19 του εισηγητή όλες μαζί «105-19 υπέρ». Όχι, δεν θέλετε. είναι μια ριζοσπαστική, μικρή αλλά ισχυρή μειοψηφία. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15, 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 17 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 18 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 19 κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά δεκτή. 106 υπέρ, κατά αποχές απολύτωται Προϋπολογισμή 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Δεκτό. 100 ε... Ναι, 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1,65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται, απορρίπτεται μάλλον 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 λέει ο πρόεδρος. Όχι, όχι. 47 διορθώνει του εισηγητή. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή Μήπως μπορούμε να κάνουμε όλες τις ε, τροπολογίες του εισηγητή μέχρι την 68 όχι 48 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεν μπορώ να τις ψηφίσω μαζί. 52 υπέρ. Κατά αποχές 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα μπορώ να ψηφίσω τις υπόλοιπες από κοινού. Ούτε τώρα. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ θέλετε έλεγχο για την 66 ωραία πέρας ψηφοφορίας 24-17 γίνεται δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές 173 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 177, βεβαίως. Πάμε. πέρας. Για την 177. 15 με 27 απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστή 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 180 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Είτε 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή τα 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Υπέρ. Κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος. Ποια ήταν, α, η 183. Πέρας ψηφοφορίας. 22-17 γίνεται δεκτή. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να πάρουμε όλες τις τροπολογίες του εισηγητή ομού. Ένα τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τις 3 ήτρε, 12, 13, 14 υπέρ. Κατά. Αποχές τεκτές. Τροπολογία 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1.89. Μπορούμε όλη αυτή την ομάδα από τροπολογίες του εισηγητή. Όχι, δεν μπορούμε. Θεέ μου. 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 191 190 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 82, 82 υπέρ κατά αποχέ. δεν βλέπω κανένα ψηφίζει κιόλα. Δύο προ ένα, δύο με ένα, αλλά εγκρίθηκε. 82 με φυσιολογικές συνδικές ψήφι υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή 93. υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτο 88 υπέρ κατά αποχές 88 και πάλι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1.94 υπέρ κατά αποχές απορριπτέται. Είναι 38 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από αυτό το ηρωικό εγώ έκανα λάθος σε μια τροπολογία θέλω να ξαναψηφίσουμε πάλι τροπολογία 146 ε, στην σελίδα γιατί υπήρχε λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας. Το άρθρο 3, εκεί που λέει στην πέμπτη σελίδα στο αγγλικό κείμενο, ε, άρθρο 3 παράγραφος 5 σε νέα στην 146. Συμφωνείτε να ξαναψηφίσουμε. Νομίζω ότι με την ε, μεγάλη ταχύτητα που ψηφίσαμε είπα ότι απορρίφθηκε ενώ υπήρχε μια θετική, θετική πλειοψηφία. Υπέρ της 146. Κατά. Αποχές. Έχει γίνει δεκτή λοιπόν. Και ερχόμαστε στην τελευταία ψηφοφορία για την ε, εντολή διαπραγματεύσεων ψήφι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «22 προς 19 και με μία αποχή γίνεται δεκτή». Σας ευχαριστώ. και χαιρετίζω τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Νέας Ζηλανδίας που είναι παρόν μεταξύ μας. Καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Es sind dabei die folgenden Mitglieder des äh, Parlaments. Επίση τα εξή μέλη του Κοινοβουλίου, Μελίσσα Λί, Ερίαν Φέλντεν, Τέλσο Ρόκεν, Γκάρι Χούτ. Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. glaube, wir haben mit Neuseeland in vielen Fragen Έχουμε κοινέ απόψει σε πολλά θέματα με την Νέα Ζηλανδία. Μα ενδιαφέρει η δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Και έχουμε και άλλα κοινά συμφέροντα. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία μαζί σα. Είχαμε κάποιε δυσκολίε στην αγροτική πολιτική ενίοτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συνεργασία στου άλλου τομεί. Σα ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σα. Έρχομαι στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης και από ό,τι γνωρίζουμε η Επιτροπή ε, συμφώνησε για να υπογραφεί η Συμφωνία Διευκόλυνσης Προξενικών Θεωρήσεων με την Ουκρανία και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ το Γενικό Διευθυντή από την Υπηρεσία του Ασύλου και της Μετανάστευσης, ο οποίος μπορεί να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση για την κατάσταση των πραγμάτων σε σχέση με το θέμα αυτό. Θα ήθελα φυσικά εν καιρό να μπορούμε να έχουμε, ή δυνατόν σήμερα ή αύριο, να έχουμε το κείμενο της συμφωνίας που έχει υπογραφεί. Κυρία Σίγρα, αν έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, καλησπέρα σε όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να πω δύο λόγια για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να σας ενημερώσω πρώτα απ' όλα ότι η Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις για την υπογραφή και την κατάληξη σε μια συμφωνία που τροποποιεί την σημερινή συμφωνία διευκόλυνσης βίζα που ισχύει τώρα στις 5 Ιουλίου. Γνωρίζω, όλοι γνωρίζουμε, τις ανησυχίες που εκφράσατε ορισμένοι από εσά στις συζητήσεις για το κατά πόσο η ολοκλήρωση της τροποποιημένης αυτής συμφωνίας είναι ότι καλύτερο κάτω από τις σημερινές πολιτικές ε, καταστάσεις και εκφράσατε κάποιες ανησυχίες για την τήρηση του κράτους δικαίου και των ε, δημοκρατικών αρχών στην Ουκρανία. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε πεπισμένοι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή, η τροποποιημένη συμφωνία. Διότι θα στείλει μήνυμα στήριξη στην κοινωνία της Ουκρανίας. Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε αυτές τις συγκεκριμένε πολιτικές ε, συνθήκες. Η τροποποιημένη συμφωνία ουσιαστικά θα ενισχύσει τις επαφές και θα ενισχύσει και τις υπάρχουσες διαδικασίες έτσι όπως έχουν σήμερα. Θα σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα ε, προσπαθώντας να αναφερθώ σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες θεωρήσεων. Έχουμε πρώτα απ' όλα από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε επίσης το θέμα ε, της διευκόλυνσης θεωρήσεων για τους δημοσιογράφους. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα ε, πολύ μεγάλη, για τα οποία μάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία η τροποποίηση της συμφωνίας. Θεσμικά μιλώντας πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντολή να διαπραγματευτεί την συμφωνία αυτή. Εμείς ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις και σας παρουσιάζουμε το σχέδιο συμφωνίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο προκειμένου να το συζητήσετε και να καταλήξετε. Τέλος, θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε, να δώσετε την συμφωνία σας, δηλαδή στην τροποποιημένη αυτή συμφωνία. Ελπίζουμε ότι θα το κάνετε αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα δώσετε δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη σας. Από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε σχετικά με τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, αυθόρμητα, θέλω να πω το εξή. Μπορώ να φανταστώ ποιο είναι το μήνυμα. Όμως η πολιτική στήριξη στην κοινωνία των πολιτών ε, πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που θα το εκλάβει διαφορετικά η κυβέρνηση τώρα παραμονέ εκλογών. Θα πει, α, κοιτάξτε, εμείς καταφέραμε να έχουμε περισσότερη ελευθερία στο σύστημα θεωρήσεων για του πολίτε μα. Είδατε τι καλά που τα κάνουμε. Λοιπόν, ναι, μεν θέλω την ελευθερία θεωρήσεων για τους Ουκρανούς βεβαίως, αλλά ανησυχώ όσον αφορά το πολιτικό μήνυμα. Είναι ένα θέμα και συγκεκριμένη στιγμή. Ακριβώς πριν από τις εκλογές δεν είμαι σίγουρος μάλιστα ότι οι εκλογές αυτές θα είναι απόλυτα σωστές και δίκες, οπότε να στέλνουμε ένα τέτοιο μήνυμα δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική ίσως και τα μέσα ενημέρωσης θα το κλάβουν διαφορετικά, θα πάει σε βάρος της αντιπολίτευσης εκεί, γιατί το μήνυμα που θα περάσουν είναι ότι κοιτάξτε εμείς είμαστε επιτυχείς όσον αφορά την πολιτική μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις εκλογές, όπως έχω πει και πριν, δεν θα ήμουν κατά. Μάλιστα θα έλεγα ναι να ισχύσει και για ολόκληρο τον πληθυσμό, αλλά να στείλουμε τώρα ένα μήνυμα νομίζω ότι θα τύχει κατάχρηση εκεί το μήνυμά μας και δεν θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ουσιώδη ζήτημα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για τις σχέσεις μας με την Ουκρανία σε όλα τα επίπεδα. Εν μέρη θα αναφερθώ στο θέμα αυτό καθευτό και μετά θα αναφερθώ και σε αυτά που είπε ο κύριος Γκάλερ πριν από λίγο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα. Έχουμε εκφράσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη θέση μας σχετικά με τα προβλήματα της δημοκρατίας στην Ουκρανία πολλές φορές με διάφορα ψηφίσματα. Το δεύτερο είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, το καθεστώς στην Ουκρανία σήμερα, σχετικά με το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γκάλερ, έτσι κι αλλιώς υπέστη κυρώσεις, μια που πάγωσε η διαδικασία σύνδεσης και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που είχε ετοιμαστεί, αλλά δεν μονογράφηκε τελικά. Το να χρησιμοποιούμε την πολιτική αυτή του καρότου και του μαστίγιου, προσοχή πώς θα εφαρμοστεί. Πρέπει να εφαρμοστεί ισορροπημένα. Αν χρησιμοποιούμε περισσότερο το μαστίγιο, καταλαβαίνω ότι είναι σε βάρος του πληθυσμού εκεί τελικά. Γιατί υποφέρουν οι πιο ευάλωτοι στην κοινωνία της Ουκρανίας και το πιο μεγάλο μέρος της κοινωνίας εκεί, οι νέοι, οι διανοούμενοι. Συνεπώς, το... να θέσουμε υπό τώρα το θέμα της ε, ελευθερίας ε, ε, όσον αφορά το σύστημα θεωρήσεων, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τις εκλογές. Εγώ σας παρακολούθησα πολύ ήσυχα κύριε Γκάλερ, οπότε σας παρακαλώ και εσείς τώρα να με ακούτε προσεκτικά. Γνώμη μου λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να διακοπεί το καθεστώς ε, αυτό, μη υποχρέωση θεωρήσουν δηλαδή. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ο κύριος Μπροκ ζήτησε την αναβολή. Το δίλημα φυσικά είναι πολύ βασικό. Τι κάνουμε, ακολουθούμε την προπαγάνδα που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση της Ουκρανίας που θα πει ότι ορίστε η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμωρεί τον πληθυσμό της Ουκρανίας ή θα πούμε ότι αν υπάρχει λόγος ε, για τιμωρία, εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά μπορούν οι σχέσεις μας να είναι κανονικές και προς όφελος του κρανικού λαού, τότε ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θεμελιώδης ερώτημα. Πρέπει να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι η Ουκρανία δεν είναι μια χώρα που αξίζει αυτή τη διευκόλυνση, αλλά ο λαός της Ουκρανίας το εξίζει και αυτή είναι η βασική διαφορά. Εμεί μέχρι τώρα σαν Ένωση προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε δύο παράλληλους δρόμους σε σχέση με τους γείτονες μας. Από τη μία ήμασταν αυστηροί απέναντι στις αρχές και από την άλλη δεκτικοί απέναντι στην κοινωνία. Ο κύριος Γκάλερ έχει δίκιο ότι οι εκλογές σαν αυτό σκοπός είναι κάτι το οποίο σαφώς θα πέσει θύμα θα έλεγα σαν διαδικασία κατάχρησης. Οι εκλογές αυτές έτσι και αλλιώς δεν θα είναι ελεύθερες και δεν μπορούν να είναι ελεύθερες αν οι ηγέτες αντιπολίτευσης είναι φυλακισμένοι και παραμείνουν φυλακισμένοι. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από πλευρά μα στον τομέα τη επικοινωνία, εξηγώντα ότι για τους λαούς παίρνουμε τα μέτρα αυτά και όχι για τι αρχέ. Σε πολλά έγγραφά μας τα τελευταία χρόνια έχουμε επαναλάβει ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας δεν θα πρέπει να γίνει μετά από την αντίστοιχη συμφωνία με τη Ρωσία. Η διαδικασία με τη Ρωσία έχει προχωρήσει αρκετά αντίθετα με την θέση που έχουμε εμείς εδώ. Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε όλα, όλοι τα ίδια επίπεδα με τους γειτονές μας, βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση στην Ουκρανία καταπιέζεται, καταστέλλεται, αλλά μπορεί να παρέμβει στις εκλογές, ενώ αντίθετα στην Λευκορασία και στη Ρωσία δεν μπορεί. Η πορεία λοιπόν προς τη δημοκρατία είναι θα έλεγα μία μακρά πορεία στην χώρα αυτή παρά τις προσδοκίες που γέννησε η Πορτοκαλή Επανάσταση. Πρέπει να είμαστε όμως δεκτικοί απέναντι στους Ουκρανούς, πρέπει να σταθμίσουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα και να προχωρήσουμε με το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων, εξηγώντας πως το κάνουμε προς χάρη των Ουκρανών και όχι των Ουκρανικών αρχών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη δουλειά της και την έκανε ε, καλά θα έλεγα. Συμφωνούμε με την συμφωνία αυτή. Πρόκειται για μια συμβιβαστική λύση. Θα ακολουθήσει μια συμβιβαστική διαδικασία έτσι ώστε να συνεχίσουμε να πιέζουμε τις αρχές της Ουκρανίας. Θα μπορούσα να πω ότι οι αρχές αυτές να συμφωνήσω με αυτούς λέγοντας θα καταχραστούν αυτή της δυνατότητας. Από την άλλη η άρνηση από πλευρά μας να συνεχιστεί η διαδικασία ή και η απλή αναβολή της διαδικασίας αυτής θα παρανοηθεί από την κοινωνία στην Ουκρανία και θα απογοητεύσει την κοινωνία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή τη χρονική φάση βασικό συνημιλωτής μας είναι η Ουκρανική κοινωνία γιατί ασκούμε σκληρή κριτική στις Ουκρανικές αρχές και θα πρέπει να φροντίσουμε τα αισθήματα της κοινωνίας περισσότερο παρά ε, τη στρεβλή απεικόνηση των θέσεων τις οποίες εκφράζει, ή, τις οποίες χρησιμοποιεί μάλλον ε, η Ουκρανική κυβέρνηση. Εγώ δεν αρνούμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκάλε. Πρέπει να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι είναι έτοιμη η συμφωνία, ότι η προοπτική τους έτσι ώστε να έχουν ε, μια επιπλέον διευκόλυνση στην επαφή μαζί μας και να ταξιδεύουν εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματικότητα και ο διάλογος, ο ειλικρινής και γνήσιος διάλογος με τις ουκρανικές αρχές ε, γιατί ξέρουμε ότι πρόκειται για μια κυρίαρχη χώρα, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές αυτές. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν. Ήδη το ότι έχει υπάρξει αναβολή για την επικύρωση της εταιρικής σχέσης είναι μια πρώτη μορφή κύρωσης, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια επιπλέον κύρωση για το ίδιο πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο αν μπορώ να προσθέσω μονάχα δύο φράσεις στο θέμα αυτό. Δεν έχουμε <clears throat> πολλές ελπίδες ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια τροποποίηση της κατάστασης μετά τις εκλογές. Αναφέρομαι στη γενική κατεύθυνση προς την οποία κινείται τώρα η Ουκρανία και ανησυχούμε φυσικά αρκετά για την κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πιο σημαντικό για μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να διατηρήσουμε την επαφή με την κοινή γνώμη και με τους πολίτες της Ουκρανίας θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Γκάλερ. Πολύ σωστά. Ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες της Ουκρανίας ότι διαφωνούμε με την προοπτική της ε, φιλελευθεροποίησης για τις προξενικές θεωρήσεις. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ουσιαστικά επιλογή. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, να δεχτούμε αυτή την φιλελευθεροποίηση και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πολύ καλή προετοιμασία που έχει κάνει για αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να αντιδράσω. Γιατί πιστεύω ότι είναι υπερβολή να μιλάμε για καθεστώς στην Ουκρανία ή να λέμε ότι είναι ελεγχόμενα τα μέσα ενημέρωσης τη στιγμή που μπορεί να μην είναι τέλεια τα μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία, αλλά σίγουρα συγκρίνονται με άλλα στις διάφορες ευρωπαϊκές μας χώρες. Αν λοιπόν λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές, εντάξει. Αλλά τι αποτέλεσμα περιμένετε αν ε, το ίδιο κόμμα ή ο ίδιος συνασπισμός κερδίσει, τι θα κάνουμε πάλι, θα αναβάλουμε τη διαδικασία περιμένοντας να κερδίσει κάποιο άλλο κόμμα. Ας τα χωρίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Έχουμε ήδη κάνει πολλά, έχουμε πιέσει πολύ. Δεν ε, επικυρώσαμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, για παράδειγμα. Ε, κάνουμε κάτι για το λαό της Ουκρανίας. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε το μήνυμά μας, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι είναι κάτι που κάνουμε για το ολό της Ουκρανίας. Έπειτα η Λευκορωσία, σας υπενθυμίζω, που ορισμένοι από εσάς τώρα τη συγκρίνουν με την Ουκρανία, εκεί λοιπόν είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία των πολιτών εκεί και ότι θα ανοιχτούμε όσο γίνεται περισσότερο για τον λαό της χώρας. Ε, για την Ουκρανία νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι τα επιχειρήματα που ακούσαμε είναι λογικά Είναι σωστό αυτό που ακούσαμε για το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και ότι πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι υποφέρουν. Όμως καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στραβά και τελικά το μήνυμα που θα στείλουμε να μην είναι αυτό που θέλουμε. Μπορεί να ακουστεί εκεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να φτιάξει ένα τείχος ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι θα ζημιώσει ακόμα περισσότερο την αντιπολίτευση στην Ουκρανία. Για μένα οι θεωρήσεις έτσι κι είναι κάτι στραβό, είναι κάτι λάθος, γιατί πάντα δημιουργούν τύχη, φραγμούς. Συνεπώς δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί στην πολιτική μας. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την πολιτική μας γενικά όσον αφορά τις θεωρήσεις. Έπειτα εγώ δεν γνωρίζω καμία Κανένα στην Ουκρανία, είτε πρόκειται για την κοινωνία των πολιτών, είτε για εκκλησία, είτε για οργάνωση, δεν ξέρω κανένα, κανένα τέτοιο φορέα στην Ουκρανία που να θέλει θεωρήσεις. Συνεπώς, εφόσον κανείς δεν είναι υπέρ του τρέχοντος καθεστώτος θεωρήσεων, καλά θα κάνουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ε, που είχαμε για την Ουκρανία, είχαμε πει ότι δεν πρέπει να συνδέσουμε το θέμα των θεωρήσεων με την πολιτική κατάσταση εκεί. Αλλιώς οι Ουκρανοί εταίροι μας θα σκεφτούν ότι προσπαθούμε να τους πατρονάρουμε. Να προσθέσω και εγώ κάποια στοιχεία τα περισσότερα επιχειρήματα είναι υπέρ ακούστηκαν και είναι υπέρ της απελευθέρωσης. Να αναφερθώ σε ένα ιστορικό, σε μια παράλληλη ιστορική αναφορά. Όταν η χώρα μας πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα και θυμάμαι πόσο χρήσιμο ήταν, πόσο θετικό ήταν όταν οι αντιπολιτευόμενοι, όταν οι, οι στο καθεστώς είχαν την δυνατότητα να πηγαίνουν στη Δύση. Αυτό ακριβώς έχουν ανάγκη και οι Ουκρανοί σήμερα. Είχα πάει στο Κίεβο πριν από δύο εβδομάδες, είχα πάει σε ένα κονσέρτο ρόκο στο κέντρο της πόλης όπου βρέθηκαν κυρίως 500.000 νέοι Ουκρανοί, τραγούδησε ο Έλτον Τζον, η Κουίν, το συγκρότημα Κουίν, και ήταν τόσο ευτυχής οι Ουκρανοί που έστω και για λίγες μέρες ανήκαν σε αυτό το οποίο ονομάζουν και ονομάζουμε και εμείς Δύση. Προσθέτω λοιπόν και εγώ τη φωνή μου στην, ε, στους συναδέλφους και είμαι υπέρ ε, της ε, βελτίωσης του ανοίγματο του καθεστώτος χορήγησης θεωρήσεων προς την Ουκρανία το ταχύτερο δυνατόν γιατί έτσι θα βοηθήσουμε τους νέους, έτσι θα βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν η χώρα τους να ανοίξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επηρεάσει την πολιτική κατάσταση μπορούμε και συμφωνώ με τους συναδέλφους, μπορούμε να βάλουμε κάποια επεξήγημα, καμιά επεξήγηματική δήλωση παράλληλα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορέσει να καταχραστεί, θα έλεγα, αυτή την απόφαση πριν από τις εκλογές που αναμένονται τον μήνα Οκτώβριο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Κύριε Ζήβιτς, εγώ δεν έχω αποστείλει καμία επιστολή, απλώς έχω κάνει μια δήλωση. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανένα τρόπο να επιβάλλει κυρώσεις στον λαό της Ουκρανίας. Αρκετή καταστολή υφίσταται από, το δικό του, από τη δική του κυβέρνηση. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία όπως έχουμε διαπιστώσει και στο Στρασβούργο αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήταν μια λανθασμένη λοιπόν κίνηση από εμά όταν η αντιπολίτευση, ένα μεγάλο μέρο τη αντιπολίτευση είναι στι φυλακέ. Δεν μπορεί κανεί να μιλήσει βέβαια για ελευθερία έκφραση. Από την άλλη πλευρά όμω αληθεύει το γεγονό ότι εμεί δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσει και ποινή στου απλού ανθρώπου. Δεν πρόκειται για απελευθέρωση πλήρω τη προξενική θεωρή. Πρόκειται για διευκόλυνση και ελάφρυνση του καθεστώτο σε ορισμένου τομεί, Αυτή είναι ακριβώ η πρότασή μα ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτοί οι οποίοι θα αποκομίσουν ε, θετικά στοιχεία. Όχι οι, τα μέλη της ολιγαρχίας, όχι οι διπλωμάτες. Θα πρέπει οι απλοί άνθρωποι, οι φοιτητέ να έχουν αυτή τη διευκόλυνση. Και νομίζω ότι είμαστε ομόφωνοι για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να τους δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα στο βαθμό του δυνατού. Και θυμάμαι και από τη δική μου χώρα τι σημαίνει η ελευθερία του να ταξιδέψει κανείς και πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να έχει την εμπειρία του να συναντήσει ανθρώπους σε χώρες όπου υπάρχει ελευθερία, το πόσο σημαντικό υπήρξε αυτό να υπάρξει δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης για τον απλό πολίτη. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που είναι μεγάλη σημασία για τον απλό πολίτη και ιδίως κάτω από τέτοιες συνθήκες. Πρέπει να το υποστηρίξουμε, αλλά σας ζητώ όπως είπα από την Κομισιόν, να έχουμε το κείμενο στη διάθεσή μας, να το ελέγξουμε καλύτερα για να δούμε κατά πόσο μας δίδει αυτά τα ωφέλη αυτή η συμφωνία και αν κάνει την απαραίτητη διαφοροποίηση. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε παρά μόνο όταν δούμε το κείμενο. Γι' αυτό για πολιτικούς λόγους θα πρέπει να έχουμε το κείμενο αυτό στη διάθεσή μας το ταχύτερο δυνατό για να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται στις λεπτομέρειες. Εντάξει, μπορώ λοιπόν να κλείσω αυτό το σημείο τη μέση τη διάταξης και περνάμε στο επόμενο που αφορά τα θέματα του προπολογισμού και δίνω το λόγο στον κύριο Κόβατσοφ. Uh, uh, Περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2013, όλα τα τμήματα. Και θέλω να δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην κυρία Γιατεμάκη. Όσο γίνεται πιο σύντομα, παρακαλώ, κυρία Γιατεμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω φιλανδικά και θα είμαι όντω σύντομη. Καταρχήν, όταν τα κράτη-μέλη καλούνται να μειώσουν τις δαπάνες τους, το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Προπολογισμών όμως και το Συμβούλιο πρότεινε 10% μείωση όσον αφορά τον προπολογισμό εξωτερικών σχέσεων, που είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ο περιορισμός αυτός, η μείωση αυτή είναι πολύ μεγάλη. Προτάθηκε καταρχήν, για ποιο λόγο. Επειδή θα υπάρξει αύξηση 7% για τη συνοχή και κάποιες χώρες ζήτησαν αυτή την αύξηση, η οποία έγινε αποδεκτή. Γι' αυτό λοιπόν ο προπολογισμό για τις εξωτερικές ε, σχέσεις πρέπει να μειωθεί. Θα ήταν καλή ιδέα αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες προτεραιότητες για όλα τα τμήματα. Δεν είναι δυνατόν όμως όλα να τα πούμε προτεραιότητα, γιατί τότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει όντως να καθορίσουμε προτεραιότητες. Και γι' αυτό ακριβώς έχω διάφορες ερωτήσεις και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Πάντως, πριν αποφασίσουμε το οτιδήποτε, προτείνω να οργανώσουμε μία ακρόαση, κατά τη διάρκεια της οποίας να εξετάσουμε προσεκτικά οι περικοπές αυτές στην πράξη τι ακριβώς σημαίνουν. Υπάρχει μια πρόταση για αύξηση 0% όσον αφορά τον προπολογισμό εξωτερική δράση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων έχει ελπίσει για 5% αύξηση. Δεν ξέρω κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε και να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Δύο είναι οι αρχές. Ευελιξία, να δούμε τις προτεραιότητές μας, δηλαδή και δεύτερον, να προσπαθήσουμε να έχουμε και προτεραιότητες στους συναφείς τομείς. Πάντως, επιτρέψτε μου να ρωτήσω μερικά πράγματα. Τι ακριβώς σημαίνει εάν οι περικοπές αυτές γίνουν αποδεκτές. Ποια τμήματα αφορούν όλα αυτά. Τελικά αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε επιπτώσεις επιτόπου και σε συγκεκριμένα θέματα. Και αυτά ακριβώ είναι που θα ήθελα να ξέρω. Όταν η δίκηση για τις εξωτερικές σχέσεις, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, Κάποιος πάει από α13 σε α14 πρόκειται για 300.000 ευρώ. Ε, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με λεπτομέρειες. Διότι εδώ δεν πρόκειται για μικρά, για λίγα χρήματα και αναρωτιέμαι, είναι λογικό να προβλέπουμε κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι παράλογο. Συνεπώς, πολύ συγκεκριμένα να έχουμε συγκεκριμένους ορισμούς, να ξέρουμε δηλαδή ακριβώς ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις επιτόπου και ποιε είναι οι προτεραιότητε του Συμβουλίου και τη Επιτροπής, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι όλα προτεραιότητα. Άρα πρέπει να καταλήξουμε στις προτεραιότητέ μας. Απαντήστε μου λοιπόν σας παρακαλώ και ακόμα και αν τις απαντήσεις δεν τις ε, πάρουμε αμέσως, αν μη τι άλλο πριν καταλήξουμε εμείς τις δικές μας αποφάσεις, πρέπει να τις έχουμε αυτές τις απαντήσεις, να ξέρουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος από τις οικονομίες αυτές που προτείνονται. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μας αφορά εμάς άμεσα, μια που και εμείς αποφασίζουμε. Όταν λοιπόν αναλαμβάνουμε κάποιες δεσμεύσεις, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι και ο δημοσιονομικός αντίκτυπος Και εδώ λοιπόν θέλω περισσότερες διευκρινήσεις. Ίσως μπορούμε να μειώσουμε τις πληρωμές αντί για τις δεσμεύσεις, αντί για τις υποχρεώσεις δηλαδή. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Σκιώδες εισηγητές τώρα. Μιχαλ Γκάλερ πρώτα. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τις ε, προτάσεις που έχει στην γνωμοδότηση της κυρία Γιάχτε Μάχη. Μίλησε για συνέργειες, για μια σειρά επίσης γενικά δημοσιονομικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προκύπτει από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης κάποια συνέργεια. Είναι και η απάντηση στην προηγούμενη κατάσταση στο ότι δεν μπορούμε μεμονωμένοι να εργαστούμε τόσο αποτελεσματικά και ότι πρέπει κάπως να συνενώσουμε τις προσπαθίες μας και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε περισσότερα εγχειρήματα σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αυτό σημαίνει και εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος μας, να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες συνέργεια στις δομέ που έχουμε δημιουργήσει και α προσπαθήσουμε έτσι να υπάρξει η πιο αποτελεσματική δυνατή εφαρμογή αυτής της ε, συνένωση προσπαθειών εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποια σημεία που εμφανίζονται κατ' επανάληψη. Παραδείγματο χάρη τα 170 εκατομμύρια η περικοπή στον τομέα 4 Εγώ εδώ δεν συμφωνώ ιδιαίτερα αν δεν υπάρξει μια μεγαλύτερη διευκρίνηση σε σχέση με τις πιστώσεις πυλωμών, οι οποίες ε, έχουν μειωθεί κατά 17% σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν όταν αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τις διαπραγματεύσεις που εμείς έχουμε αποφασίσει να έχουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερη λογική εκεί. Επίσης το μέσο ε, έχουμε περικοπές λιγότερες προς τα, για τις νότιες χώρες γειτονίας και περισσότερο για τις ανατολικές χώρες. Επίσης σε σχέση με την Παλαιστίνη παραμένει εκεί πέρα ένα ποσό σταθερό για τη δέσμευση υποχρεώσεων όπως πρότεινε η Κομισιόν αλλά δεν είναι επαρκή αυτά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Επίσης για το προενταξιακό μέσο υπάρχουν κάποιες περικοπές για τη μεταβατική, μεταβατική δημιουργία δημοκρατικών θεσμών σε ορισμένες υποψήφιες χώρες και εκεί είναι μικρότερο το ποσό από την πρόταση της Κομισιόν Έχουμε 18 εκατομμύρια τα οποία μειώνται στις πιστώσεις πληρωμών για τις υποψήφιες χώρες. Το μέσο σταθερότητος επίσης θεωρώ δεν θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι μειώνονται και εκεί οι χρηματοδοτήσει, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επωφελώ και πιστεύω και εκεί δεν είναι ευτυχέ το γεγονός ότι περιορίζονται τα κονδύλια. Αυτά θα ήθελα να πω. Now for the Οι πολιτικές ομάδες τώρα έχουν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου πολιτική ομάδα συμφωνούμε ιδιαίτερα με την γενική κατεύθυνση που έχει αναφέρει ο κύριος Γκάλερ. Θεωρούμε ότι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια σειρά από στόχου για τους οποίους νομίζω ότι εν γέννη συμφωνούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε του στόχου των συνδικών σε ό,τι αφορά την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη συνεργασία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιστήσουμε στόχους ανάπτυξη, διεθνέ εμπόριο, όλα αυτά. Επομένως, ο προπολογισμό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα άγχος, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο επίτευξη των στόχων μα. Νομίζω λοιπόν ότι και η συγγήτρια του προπολογισμού κατανοεί ότι ο προπολογισμό του 2013 είναι ένα κομβικό προπολογισμό, ο οποίο θα σηματοδοτήσει και την πορεία των δημοσιονομικών προοπτικών για το μέλλον. Μας φαίνεται πάρα πολύ ανησυχητικό το να βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απογυμνώνεται από το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει σε διεθνές επίπεδο. Η Κομισιόν θέλει να αυξήσει τον προϋπολογισμό κατά 5% σε σχέση με το 2012. Αυτό είναι θετικό γιατί η Κομισιόν έχει την καλύτερη γνώση του κόστους των πολιτικών που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και μας φαίνεται ότι θα είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού ε, και το τι σημαίνει για κάθε γραμμή το 5 αυτό το 100. Το Συμβούλιο θέλει να περικόψει 171 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 171 εκατομμύρια από τα οποία 37 παραδείγματος χάρη είναι σε πιστώσεις πληρωμών για την πολιτική γειτονία με τις μεσογειακές χώρες. Αυτό μας φαίνεται πολύ σοβαρό. 8 εκατομμύρια ευρώ περικόπτονται στη συνεργασία για την ανάπτυξη. 38 εκατομμύρια για το περιβάλλον και την προστασία των φυσικών πόρων και αυτό περιλαμβάνει και τους ενεργειακούς πόρους. Ή δύο λιγότερα εκατομμύρια για την ισότητα των φύλων. Όλα αυτά αποστερούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να φέρει σε πέρα μια σειρά από πολιτικέ που δεν είναι απλώ ε, μια πολυτέλεια ή ένα καπρίσιο, αλλά είναι πολιτικέ τι οποίε θέλουμε εμεί να υλοποιήσουμε γιατί αποτελούν του στόχου μα. Γι' αυτό εμεί δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την αρχική προσέγγιση του Συμβουλίου βάσει του ε, εγγράφου αυτού που έχουμε από την 5η Ιουνίου, αλλά δεν έχει ακόμα επίσημο χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν τα 563 εκατομμύρια για το περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μας, ξέρουμε ότι αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για τις ε, πολιτικές που προανέφερα. Υπήρξε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για να χρηματοδοτήσουμε τους τομείς προτεραιότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αυτό και φέτος, να έχουμε μια, ένα επακριβή καθορισμό των προτεραιοτήτων Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται 300 εκατομμύρια για να διατηρήσουμε μερικούς ζωτικούς τομείς και δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στα σημεία αυτά Ξέρουμε ότι ο προπολογισμό είναι πάντα ένα σημείο τριβή μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων. Δεν θέλουμε να είμαστε δημαγωγικοί σε σχέση με του ε, πόρου που θέλουμε να δώσουμε στι ορισμένε πολιτικέ, αλλά θέλουμε να είμαστε λογικοί. Κυρία Λέζινγκ, από την ομάδα των, ε, της σα σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας μου και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση από την κυρία Γιάχτε Μάχη και συμμεριζόμαστε σε ε, πολλά σημεία την έμφαση που έχει δώσει η συγήτρια στα θέματα εξωτερικής πολιτικής για το 2013. Βλέπουμε επίσης ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση για να επιτευχθεί η λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική ανεξαρτησία των οντοτήτων και των χωρών που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θεωρούμε ως ΓΚΟΕ ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η κοινοβουλευτική διάσταση στα θέματα αυτά συνεργασίας και αυτό θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα περιληφθεί στον ε, προϋπολογισμό και θα ήθελα εδώ να ξέρω ποια είναι η άποψη της Κομισιόν. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα που έθεσε η κυρία εισηγήτρια σε σχέση με τις ενδεχόμενες συνέργειες και εξοικονομήσεις που ανέφερε και ο κύριος Γκάλερ σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εγώ είμαι κάπως σκεπτικιστική σε σχέση με τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν απτές εξοικονομήσεις σε επίπεδο κόστους και σίγουρα αυτή η συνέργεια δεν πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος της δημοκρατίας γιατί αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο να συμβεί στον τομέα της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης. Εκπρόσωπος ο κύριος Μπούσερ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αρχίσω από τη δεύτερη ερώτηση της εισηγήτριας. Πράγματι, η υπηρεσία μα ε, ζητάει 10 θεσει α α13 να γίνουν α14, κάτι το οποίο απορρέει από την εφαρμογή του καταστατικού που διέπει του υπαλλήλου, που προβλέπει ένα ποσοστό προαγωγής κάθε χρόνο για κάθε συγκεκριμένο βαθμό. Υπολογίσαμε λοιπόν για τον κάθε βαθμό τις προγωγές που αντιστοιχούν στο ποσοστό που προβλέπετε, αν ε, τη συγκρίνουμε βέβαια και από τις κενές θέσεις και διαπιστώνουμε ότι στο βαθμό α14 υπάρχει ένα έλλειμμα για πραγωγή από τους, 10, από τους α13. Και γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε να γίνουν οι προαγωγές αυτές. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε πολλούς υπαλλήλους στο βαθμό α13 είναι ότι ήρθανε πάρα πολλοί υπάλληλοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τους κληρονομήσαμε κατά κάποιο τρόπο εμείς στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν πρόκειται για προσλήψεις που έγιναν από τα κράτη-μέλη. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η Α13 δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή η πραγωγή, αλλά το προβλέπει το καθεστώς. Και αν δεν γίνει, τότε θα υπάρξουν ε, περισσότερες κενές θέσεις στο α13, οπότε θα πρέπει να ε, πάρουν προαγωγή λιγότερη α12 και ε, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία, λιγότερους α11 να προάγουμε στην α12 και ούτω καθεξής. Άρα ολόκληρη η πυραμίδα θα υποφέρει αν δεν γίνουν οι προαγωγές αυτές. Θέλουμε να εφαρμόσουμε εμεί όμως το καθεστώς γιατί πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Ε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα άλλα όργανα τα οποία επίσης ε, κάνουν προαγωγές και δεν θα έπρεπε να τις κάνουν πιο γρήγορα από ότι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε να γίνει η προαγωγή αυτή. Το κόστος δεν είναι τόσο πολύ, είναι κάτω από 200.000 όταν μιλάμε για 500 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον προπολογισμό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσοστό δεν πρόκειται να αλλάξει ε, με σημαντικό τρόπο το σύνολο του προπολογισμού. Τώρα, για το άλλο ερώτημα. Τι θα κάνουμε εμείς με τη θέση του Συμβουλίου. 0% 2013. Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα. Γιατί πέρυσι είχε γίνει συμφωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να προβλέψουμε ήδη περικοπές 1,3% σε σχέση με το 2012 προς το παρόν. Οι περικοπές αυτές ήρθαν από κονδύλια που είχαν παγώσει για αποστολές που μειώθηκαν κατά 10% το 2012. Παγώνουν λοιπόν το 2013. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να βρούμε τρόπο να κάνουμε περισσότερες περικοπές. Θα μπορούσαμε να απαρατηθούμε από τις 20 θέσεις για τις αντιπροσωπείες ή για άλλες 20 θέσεις που προβλέπονταν το 2012 με πιστώσεις για τρεις μήνες να μην συνεχιστούν. αν πληρώσουμε για 12 μήνες αντί για 3 μήνες, 1% είναι η αύξηση του προπολογισμού της υπηρεσίας μας. 1% δηλαδή την οικονομία που θα κάνουμε. Βέβαια έτσι δεν ενισχύονται οι αντιπροσωπείες με τις θέσεις αυτές που προβλέπονται. Εξάλλου προβλέπονται από το 2012. Ένα δεύτερο θέμα τώρα κάπου αλλού δηλαδή που θα μπορούσαμε να κάνουμε οικονομία, είναι κάποια έργα για τη, κάποιες για την ασφάλεια, κάποια θέματα ασφάλειας που έχουμε, για το Ιράκ πρώτα απ' όλα. Δυνάμεις που πρέπει να φύγουν από το Ιράκ. Χρειάζεται όμως να φροντίσουμε για την προστασία και την ασφάλεια εκεί. Το ίδιο και για το Αφγανιστάν, όπως επίσης και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας ε, της αντιπροσωπείας μας εκεί και κρατών μελών που βρίσκονται εκεί. Τέτοια έργα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια θα μπορούσαν να μην γίνουν. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την παρουσία γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που δεν ξέρω πώς να λύσω. είχαμε πάντα περισσότερους υπαλλήλου από τις πιστώσεις που προβλέπονται στον προπολογισμό σε αυτή την περίπτωση. Το Συμβούλιο το 2013 θέλει να δώσει χαμηλότερες πιστώσεις από το 2012. Θα έπρεπε να γίνει κάποια διάκριση του προσωπικού που είναι με σύμβαση. Δεδομένου λοιπόν ότι Πρόκειται για χώρες όπου υπάρχει αύξηση μισθών, πληθωρισμός και αυτό επηρεάζει το αποτέλεσμα. Έχουμε επίσης πρόβλημα και για το ενίκιο της έδρας. Θα μπορούσαμε να κόψουμε 2 εκατομμύρια. Κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί από τις συμβάσει για τα νέα κτίρια της υπηρεσίας μας, που εγκρίθηκαν όμως πρόσφατα από τις αρχές επί του προπολογισμού και υπάρχει και σύμβαση για το κτίριο Κόρτεβερκ. Δύο εκατομμύρια λοιπόν, αν δεν τα έχουμε, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ε, πληρώσουμε για τη σύμβαση. Στις χώρες που είμαστε κατεστημένοι, έτσι κι αλλιώς υπάρχει κάποια αύξηση στα νίκια, οπότε δεν βλέπω πώς θα πληρώσουμε τελικά τα ενίκια για τις αντιπροσωπείες μας που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, δεν θα σας τα παριθμίσω όλα, αλλά πάντως είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε λύσει μέχρι σήμερα. Θέλω να πιστήσω επίση την προσοχή σας ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης εξαρτάται και από τις τη συλλαγματική ε, κατάσταση, τις ισοτιμίες. Όταν γίνονται μεγάλες πληρωμές σε άλλα νομίσματα, υπάρχει μια αύξηση για την αλληλεγγύη. Όταν το ευρώ από 1,40 που ήταν κατά μέσο το 2011 πάει στο 1,30 που ήταν στα τέλη Μαΐου του 2012, εμείς χάνουμε 500.000 το μήνα. Και αν συνεχίσει να μειώνεται στο 1,25 που είναι τώρα, χάνουμε επιπλέον 150.000 το μήνα. Αν λοιπόν έχουμε έναν πολύ περιορισμένο προπολογισμό, καταλαβαίνετε, έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα, δεν μπορούμε δηλαδή να απορροφήσουμε τι αλλαγέ στην ισοτιμία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε. Γι' αυτό και θέλαμε μια αύξηση στην ε, συνδιαλλαγή πάνω από το ποσοστό του 0% γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας και να τις συνεχίσουμε να τις καλύπτουμε στα επίπεδα που ήταν το 2012 αλλά θα αναγκαστούμε να, κάνουμε, να αποχωριστούμε προσωπικό το οποίο μας ήταν απαραίτητο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπέρσε. Πολλά είπατε τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ο εισηγητής θα το κάνει. Και μιας και δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση για την, κατάθεση για, τις... για την προθεσμία κατάθεση ε, τροπολογιών. 16 Ιουλίου, απογευματινή για τις τροπολογίες που τροποποιούν τις θέσεις του Συμβουλίου σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού για την έκθεση για τεμάκι. Η γραμματεία είναι στη διάθεσή σας για τα μέσα κατάθεσης των τροπολογιών αυτών. Το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών. Γι' αυτό παρακαλώ θα διακόψουμε για λίγα λεπτά.